Και βέβαια, αυτό δεν ήταν καθόλου τυχαίο. Η ισότητα ανδρών και γυναικών, μολονότι πρέπει να αποτελεί μια σημαντικότατη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι κάτι το οποίο δεν τηρείται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να καταφέρουμε να προασπίσουμε την αρχή αυτή. Όταν χτυπάμε γυναίκες, ουσιαστικά χτυπάμε κάτι το οποίο αποτελεί σημαντικότατη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ήθελα να πω ότι βρισκόμαστε στο πλάι των συγγενών και των οικογενειών των δύο αυτών γυναικών που δολοφονήθηκαν χθε στη Μασαλία εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας προς τη γαλλική αυτή και ευρωπαϊκή πόλη και εκφράζουμε όλο και περισσότερο την αποφασιστικότητά μας να προασπίσουμε τις αρχές τις οποίες, τις οποίες πιστεύουμε. Δεν πρόκειται να αλλάξουμε τον τρόπο ζωή μας, δεν πρόκειται να λειτουργήσουμε διαφορετικά, θα συνεχίσουμε να καταπολεμούμε τρομοκρατία. Πριν από μερικά λεπτά μέσω μιας ανακοίνωσης το Ισλαμικό κράτος ανέλαβε την ευθύνη της τρομοκρατικής επίθεσης που έλαβε χώρα στο Λας Βέγγας. Ουδής δεν μπορεί να καταλάβει πώς μπορεί ένας άνθρωπος να πάρει την απόφαση να προχωρήσει σε τόσο αιματηρές επιθέσεις εναντίον άλλων ανθρώπων. Σε κάθε περίπτωση οποιοδήποτε κι αν είναι ο λόγο, γιατί μέχρι στιγμή ακόμα οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν έχουν επικυρώσει ότι όντω πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση, πάλι εμεί ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ω Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζουμε την αλληλεγγύη μα και τα ειλικρινή μα συλληπιτήρια προ όλου εκείνου που ενεπλάκησαν προς την, στα πλαίσια της ματηρής αυτής επίθεση. Βρισκόμαστε πάλι στο πλάι των συγγενών και των οικογενειών των θυμάτων που χάσανε ουσιαστικά τους δικούς τους σε τέτοιες δραματικές συνθήκες. Και πάλι ευχαριστούμε τις αρχές εκείνες οι οποίες έδρασαν αμέσως προκειμένου να βοηθήσουν τους υπόλοιπους πολίτες. Επίσης το Σάββατο στο Έτμοτον του Καναδά έλαβε χώρα μια άλλη τρομοκρατική επίθεση και για αυτήν λοιπόν και για τις υπόλοιπες δύο θα ήθελα να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή. Κυρίσω την επανάληψη της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είχε διακοπήσει στις 14 Σεπτεμβρίου 2017. Τα συνοπτικά πρακτικά της 14 Σεπτεμβρίου 2017 και τα κείμενα που εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίες αυτή έχουν διανεμηθεί. Υπάρχουν παρατηρήσεις. Τα συνοπτικά